και ισπανικά, θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα τα ελληνικά. Του σχεδίου ημερησία διάταξη δεν έχουμε αντιρρήσει, οπότε το σχέδιο τη ημερησία διάταξη εγκρίνεται. Το δεύτερο είναι η έγκριση των πρακτικών. Τα πρακτικά διαβάστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε θεωρούνται εγκριθέντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγες μέρες οι Ισραηλινές αρχές ενέκριναν σχέδια για την κατασκευή σχεδόν 2.000 οικιστικών μονάδων στη Δυτική Όχθη. Ταυτόχρονα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έκρινε ότι το κράτος μπορεί να κατεδαφίσει τα σπίτια της Παλαιστινιακής κοινότητας Χαν Αλάχμα στη ζώνη γάμμα των κατεχομένων παραστατικών εδαφών και να μεταφέρει του κατοίκου από τα σπίτια του σε άλλη τοποθεσία. Πρέπει να πω αυτόν τον οικισμό τον έχουν επισκεφθεί η αντιπροσωπεία μα. Έχουμε κάνει πάρα πολλέ φορέ παραστάσει ενάντια σε αυτήν την κατεδάφιση ε, του, του οικισμού και να πω ότι στην κοινότητα μάλιστα λειτουργά και ε, νηπιαγωγείο το οποίο ε, χτίστηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμεί συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη λύση δύο κρατών και τι ελπίδε για μόνιμη ειρήνη και το απόθεμα γη για ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτο με εδαφική συνέχεια. Και ακριβώ αυτό πρέπει, έχει ξεκινήσει και με ένα συστηματικό οργανωμένο τρόπο να μην υπάρχει αυτή η εδαφική συνέχεια. Ε, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και οι πολιτικέ από τη μια επέκταση των οικισμών και από την άλλη η κατεδάφιση ε, ε, των οικισμών των Βεδιούνων αλλά και άλλων οικισμών. Ε, είναι σαφές ότι με την επέκταση των οικισμών κάτι που το διεθνές δίκαιο ορίζει ως παράνομο το Ισραήλ εδραιώνει μια πραγματικότητα στην οποία υπάρχει ένα μόνο κράτο με άνισα δικαιώματα, μόνιμη κατοχή και συγκρούσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι δηλώσει μας δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο οι αναγκαστικέ εκτοπίσει, εξώσει, καταφύσει και κατασχέσει Παλαιστινιακών σπιτιών συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά ανοιχτά και έντονα για τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνού δικαίου. Ωστόσο, το Ισραήλ μα αγνοεί, γιατί θεωρεί ότι δεν διαδραματίζουμε τον ουσιαστικό ρόλο και γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε μια διαφορετική γλώσσα για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Μια γλώσσα που θα κάνει το Ισραήλ να αντιστρέψει την επικιστική πολιτική επέκτασή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ και βάσει τη ζωή αυτή μπορεί και πρέπει να ασκήσει εξουσία. Πρέπει να διασφαλίσουμε, για παράδειγμα, ότι τα προϊόντα που προέρχονται από του εν λόγω οικισμού δεν επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα που ισχύουν για τα, για τα προϊόντα που προέρχονται από το ίδιο το Ισραήλ βάσει τη Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ισραήλ. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε και πέρα από αυτό. Θα θυμάστε την έγκριση των κατευθυντήρων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον οικισμό το 2013 και τη μόχλευση που δημιούργησε σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στο ερευνητικό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Την εποχή εκείνη το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ως αντίδραση στις κατευθυντήριες γραμμές. Εν τέλει τα πράγματα άλλαξαν όταν η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ισραήλ άσκησε πίεση στι αρχέ επειδή έκρινε ότι η αποχώρηση από το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 θα αποτελούσε ένα μεγάλο πλήγμα. Το ίδιο θα μπορούσε να υποθεί και για την πολιτική μια αναγνώριση τη Ισραηλινή κτηνιατρική επίβλεψη πέραν από την πράσινη γραμμή, η οποία ουσιαστικά απαγόρευε την εισαγωγή βιολογικών και ζωγιών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκμεταλλεύσει όπου εκτρέφονται κοτόπουλα αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν διαφορετικέ γραμμέ παραγωγή για τα κοτόπουλα που εκτρέφονται στου χειρισμού και για εκείνα που εκτρέφονται εντό τη πράσινη γραμμή. Δεν πρέπει να αστιάζουμε μόνο στου οικισμού, αλλά και στι κρατικέ και χρηματιστηριακέ οντότητε που στηρίζουν την κατασκευή των οικισμών. Ίσως αυτό να είναι ο μόνο τρόπο να αναγκαστεί το Ισραήλ να προβεί σε μια συζήτηση γύρω από τα θέματα των επικισμών. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα για την τήρηση του διεθνού δικαίου και δεν θα πρέπει να διστάζουμε να διερευνήσουμε τέτοιε επιλογέ. Από τι σημερινέ ανακοινώσει δεν θα μπορούσε να λείψει η αναφορά μου στην έκτακτη συνεδρία τη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ που έγινε την περασμένη εβδομάδα, όπου ενέκρινε ψήφισμα το οποίο προβλέπει διεθνή προστασία στον Παλαιστινιακό λαό. Παρά τι σφοδρέ πιέσει και εκβιασμού που ασκούσαν επί μέρε ΗΠΑ, 120 κράτη του κόσμου στήριξαν το ψήφισμα, μόλι μόνο 8 το καταψήφισαν, ενώ 45 κράτη τήρησαν αποχή. Το ψήφισμα, παρότι μη δεσμευτικό νομικά, καλεί το Γενικό Γραμματέα του ΕΕ να υποβάλει εντό 60 ημερών έκθεση και να παρουσιάσει προτάσει για τη δημιουργία ενό μηχανισμού για τη διεθνή προστασία των αμάχων Παλαιστινίων στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένη τη λωρίδα τη Γάζα και τη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ζητά ακόμα να αφηθεί το προσωπικό ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια να επιτοπελέσει το έργο του απρόσκοπτα. Το ψήφισμα, όπω υπέδειξε ο εκπρόσωπο τη Παλαιστίνη, εδράζεται στο διεθνέ δίκαιο συμπεριλαμβανομένου του Διεθνού Ανθρωπιστικού Δικαίου αλλά και σε όλα τα σχετικά ψήφισμα του ΟΕ για τον Παλαιστινιακό. Περιλαμβάνει μάλιστα αναφορέ καταδίκη στην υπερβολική και διάκριτη χρήση βία από τι Ισραηλινέ δυνάμει ενάντια σε αμάχου Παλαιστινίου, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και ιατρικού προσωπικού, ενώ καλεί το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τι διεθνεί συμβάσει για την προστασία των αμάχων εν καιρό πολέμου. Το ψήφισμα αυτό ήρθε ω απάντηση στο μπλοκάρισμα ενό αντίστοιχου αλλά νομικά δεσμευτικού ψηφίσματο που είχε προταθεί από το Κουβέιτ στη συζήτηση τη 1η Ιουνίου 2018 στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ, όπου η άσκησα βέτο. Η αντιπροσωπεία μα χαιρετίζει το ψήφισμα, ανεξάρτητα αν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν χωρισμένα. Ε, περίπου τα μισά ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματο, τα άλλα μισά τήρησαν αποχή. Εν τούτης εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό ψήφισμα και αναμένουμε από τη διεθνή κοινότητα να λάβει δράση για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού, ο οποίο για δεκαετίε αγωνίζεται αδιάλειπτα για τη δημιουργία ενό κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτου στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έχω καλωσορίσει στην αρχή τον Χάου Λόβατ, επιστημονικό συνεργάτη και συντονιστή του όργου Ισραήλ Παλαιστίνη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, ο οποίο θα μα βοηθήσει να ανοίξουμε εκ νέου τη συζήτηση σήμερα. Ο κύριο Ντόβατ έχει ερευνήσει ουσιαστικά το θέμα και έχει γράψει πολλά για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη διαφοροποίηση, την αλλά και του Ισραηλού οικισμού. Ασχολείται για πάρα πολλά χρόνια γύρω από τα θέματα Ισραήλ-Παλαιστίνη και ε, θεωρώ ότι με την παρέμβασή του θα φωτίσει πτυχέ που μα ενδιαφέρουν και ε, έτσι ανοίγω τη συζήτηση δίνοντας το λόγο στον κύριο Λόβατ για να καταθέσει την εισήγησή του. Ο λόγος σε σένα. Thank Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για να μιλήσω για το θέμα. Να ξεκινήσω με μια ζωφερή εικόνα, απεσιόδοξη, κλασική για τέτοιες συζητήσεις δεν υπάρχει τίποτα καινούριο σε αυτές τις αξιολογήσεις δυστυχώς. Όπως ε, είπε και η ίδια η ύπατη εκπρόσωπος, με την πορεία τη σημερινή θα οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα και μόνο. Αν δεν είναι ένα κράτος, δύο κράτη μάλλον, θα έχουμε ένα κράτος ε, με άνισα δικαιώματα για τους Παλαιστινίους. Το θέμα είναι πότε θα γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα, μήπως έχει ήδη γίνει, υπάρχει μια συζήτηση γι' αυτό, αλλά δυστυχώς προς τα εκεί κατευθυνόμαστε και για να είμαστε δίκαιοι, αυτοί που είναι εντός του Ισραήλ, κυρίως ε, η κυβέρνηση, το κίνημα των ε, οικισμών, αλλά και όλοι οι πολιτικοί υποστηριχτέ ε, πιέζουν για να φύγει το θέμα του Παλαιστινιακού από το τραπέζι. Τις γραμμές του 1967 να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Και κερδίζει αυτό το στρατόπεδο. Δεν σημαίνει αυτό ότι τελειώνει αυτή η συζήτηση. Θα υπάρξουν και νέε πραγματικότητε που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαφορετική κατάσταση, μια άλλη νοοτροπία που θα απαιτήσει ακόμα πιο δύσκολε συζητήσει, όχι μόνο από πλευρά Ισραήλ και Παλαιστίνη, αλλά και για του Ευρωπαίου πολιτικού. Αν σκεφτούμε για το πώ θα υπεραπιστούμε τη λύση των δύο κρατών, ε, τότε φαντάζομαι, που και πόσο δύσκολο είναι, φανταστείτε όταν αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα ως έχει. Ή όταν αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη apartheid ή άλλε τέτοιε σκληρέ προτάσει για να αναγκαστούμε να περιγράψουμε την πραγματικότητα. Όταν φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, όταν υπάρξει αναγνώριση αυτή, τότε θα έχουμε κάποιε δυνατότητε. Καταρχά, το κίνημα απελευθέρωση τη Παλαιστίνη κάποια στιγμή ε, δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ε, υπό τον πρόεδρο Αμπάς, αλλά υπό τον διάδοχό του κάποια στιγμή θα υπάρξει μια Παλαιστινιακή ηγεσία που θα πει αρκετά ως εδώ. Γιατί θα πρέπει η συνέχεια να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο αυτό της λύσης ε, των δύο κρατών, αφού δεν υπάρχει πρόοδος, όλα οδηγούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και τότε θα προκύψει μια νέα Παλαιστινιακή στρατηγική, είτε θα ζητήσει μέσα σε ένα κράτος ίσα δικαιώματα, ε, πολιτικά δικαιώματα, με την χρήση βίας. Δεν ξέρουμε τι θα δείξει το μέλλον. Αυτό είναι πάντως μια πιθανότητα. Μια άλλη εναλλακτική είναι, εάν ε, υπάρξει μια πιο αποφασιστική διεθνή κοινότητα και δεδομένη τη κατάσταση τη διεθνού κοινότητα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά για την ε, γενικότερη υπεράσπιση τη συνταγματική και διεθνού τάξη, και αν υπάρξει μια διεθνής κοινότητα η οποία να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο πραγματικά, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Φυσικά εδώ πρέπει να ακουστούν και επικρίσεις για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το εξή. Να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έκανε. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αδυναμίες στην ευρωπαϊκή πολιτική, και στο όραμα της Ευρώπης για το πώς θα λυθεί το, η σύγκρουση, αλλά και εσωτερικές διαρρέσεις στην Ευρώπη και χάσματα ανάμεσα στη ρητορία μας, ε, στο αφήγημά μας και στο βαθμό στον οποίο είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε και να υπρασπιστούμε τη λύση των δύο κρατών. Τούτου κλεχθέντος, νομίζω ότι είμαστε αποτελεσματικοί γιατί κρατήσαμε την ε, ίστατη γραμμή για κάποια θέματα, ας πούμε, ειδικά τώρα μετά τη διολύστηση των Αμερικανών. Και είπαμε μέχρι εδώ τουλάχιστον, δεν είπα πιο πίσω και είμαστε αποτελεσματικοί για να κρατήσουμε το θέμα ε, στους ε, προβολείς. Ε, να μιλάμε για παραβίαση του διεθνούς ε, δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ήταν έτοιμη να το στηρίξει ε, σε πολυμερή φόρουμ, στο ICC, στο Διεθνές δηλαδή Ποινικό Δικαστήριο κτλ. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, συζητάει, παρά δεν έχει κάνει κάτι άλλο, τουλάχιστον συζητάει, ε, που είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που κάνουν άλλοι Ε, υπάρχει ας πούμε άπλετο φως που έχει χυθεί για το πρόβλημα των ε, οικισμών χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ρητορία της. Και έχει κρατήσει και το θέμα του Παλαιστινιακού κράτους ε, στην επικαιρότητα, στο τραπέζι. Κάτι που αμφισβητεί όχι μόνο η Ισραηλινή κυβέρνηση, αλλά στο μέλλον <laughs> και ήδη ακόμα μπορούμε να πούμε η Αμερικανική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τραμπ. Ε, και το ότι είναι ε, αποδεκτές παράμετροι ε, διεθνώς για την επίλυση του προβλήματος και την δημιουργία ε, των δύο κρατών, τα σύνορα του 1967 και η μη κυριαρχία του Ισραήλ πάνω στους, στα κατεχόμενα και στους οικισμούς. Αυτά παρά τις αδυναμίες μας, τις εσωτερικές διαρρέσεις μας κτλ. Έχουμε, τα έχουμε κρατήσει στην επικαιρότητα. Και το βασικό εργαλείο είναι η διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αναφέρεται η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ανακεφαλαιώσω είναι διαφοροποίηση αυτή, ορισμένοι μπορεί να το ξέρετε, αλλά βασικά διαφοροποίηση είναι ένα όρος για να περιγράψουμε το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έκανε και τι κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια χοντρικά, ας πούμε, στις σχέσεις της με το Ισραήλ. Εδώ και δέκα και πλέον χρόνια ε, έχουμε βαθύτερους δεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Παρότι όμως η κατοχή δεν σταματάει και καθότι ε, επεκτείνονται οι οικισμοί, παρά τους δεσμούς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια πρόκληση. Πώς θα, αντιμετω... θα αντιμετωπίσει τους οικισμούς του Ισραήλ, στις σχέσεις της με το Ισραήλ. Πώς θα τους εντάξει, τι θα κάνει γι' αυτό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει να έχει βαθύτερες, όλο και βαθύτερες σχέσεις με το Ισραήλ αλλά αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με την επιθυμία του Ισραήλ να επεκταθεί, να επεκταθεί στο στα Παλαιστινιακά εδάφη και να βάλει τους ε, οικισμούς ε, μέσα στο κοινωνικό-οικονομικό ιστό του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, κάνει εκούσα-άκουσα όλο και περισσότερο, αλλά ε, με βάση τη δική της εσωτερική λογική, νομική λογική κάνει κάποια βήματα ούτω ώστε να αποκλείσει τους ε, οικισμούς ε, και τα προϊόντα τους και τα λοιπά από τις σχέσεις της. Έχουμε ακούσει κάποια παραδείγματα, τι σημαίνει εδώ, ας πούμε τα κοτόπουλα και τα λοιπά που ανέφερε ο πρόεδρος. Αυτό υπαγορεύεται λόγω του DNA της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως εσωτερική αγοράς που έχει τις δικές της κανονιστικές πρακτικές και τους δικούς τους νόμους, αλλά και λόγω του διεθνούς δικαίου. Και είδαμε αντίστοιχα μέτρα σε άλλες συγκρούσεις. Μερικές φορές τα εφαρμόσουμε πολύ πιο έντονα, όπως στην Κρυμαία όπου εμείς δεν αναγνωρίζουμε την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας από τη Ρωσία. Ε, μιλάμε για την κυριαρχία της ε, Κρυμαίας. Ε, και επίσης στη Δυτική Αφρική, όπου το κάνουμε λιγότερο, με λιγότερη έμφαση. Έχουμε δύο αποφάσεις σχετικές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το θέμα αυτό. Άρα δεν έχουμε αιμονή με το Ισραήλ και με την Ισραηλινή κατοχή. Δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκασμένη να το κάνει αυτό και το κάνει παρότι μερικές φορές το κάνει πραγματικά ακούσα άκουσα, δεν, δεν θέλει να το κάνει ή την αναγκάζει το δικαστήριο να το κάνει. Το κάνει παρόλα αυτά. Ε, τι είναι η διαφοροποίηση λοιπόν, όλα αυτά τα λέω για να σας πω ότι προστατεύουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος μέλος από τις ε, διεθνώς ε, παράνομε πράξει την ε, προσάρτηση εδαφών και την υπερβολική βία που απορρέει από την παρατεταμένη κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να θεωρηθεί ως νομική αναγκαιότητα, αλλά και ως αντανάκλαση της λογικής τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της νομικής τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει να προστατεύσει την ακαιρεότητα της ένωμη τάξης της. Αυτό στην πράξη τι σημαίνει. Συχνά το Ισραήλ αναγκάζεται να δεχτεί τη θέση, τη νομική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ε, συζητάει αυτά τα θέματα στις διμερείς σχέσεις, στο βαθμό που επιθυμεί να συνεχίσει αυτές τις διμερείς σχέσεις, να κάνω και κάποιες διευκρινήσεις για να σας εξηγήσω τι δεν είναι αυτή η διαφοροποίηση. Ε, είδαμε μια συντονισμένη εκστρατεία της, της Ισραηλινής κυβέρνησης ε, των υποστηριχτών ε, των οικισμών για να ανασκευάσουν το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. η διαφοροποίηση αυτή ε, γίνεται και για ηθικούς και πολιτικούς λόγους. Ή μάλλον, η διαφοροποίηση συγγνώμη, γίνεται μόνο γιατί νομικά είναι υποχρεωτικό. Ε, είναι τεχνικά τα μέτρα και όχι μόνο ηθικά. Ε, επομένως, δεν είναι κυρώσεις. Πολιτικά δεν αναγκαζόμαστε από τίποτα. Είδαμε κυρώσει εναντίον τη Ρωσία, το Ιράν κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά την είναι κύρωση. Το καταλαβαίνει κανεί αμέσω. Το να αποκλείουμε τα Ισραηλινά κοτόπουλα, ας πούμε, το να θεωρηθεί ως ως υπερβολική και μεγάλη κύρωση θα ήταν υπερβολικό. Ε, για να κάνουμε λοιπόν αυτά τα λόγια, για να κάνουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα ε, στην πολιτική διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εμποκοτάρισμα και τις κυρώσεις, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η διαφοροποίηση επίσης δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετό για να κατευνάσει τα πνεύματα των Παλαιστινίων που θα ήθελαν και μποϊκότ, μποϊκοτάρισμα και ε, κυρώσεις. Η διαφοροποίηση είναι το ελάχιστο δυνατό δηλαδή που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία περίπτωση δεν είναι το μέγιστο που μπορεί να κάνει. Έτσι. Πόρο απέχει από το μέγιστο. Τα επόμενα λοιπόν λεφτά θα πάω σε κάτι άλλο πριν πάω στις συστάσεις. Νομικά χρειάζεται η διαφοροποίηση. Αλλά ως πολιτική δεν έχει μεγάλη αξία για να για να περάσεις και να εξαναγκάσεις τους άλλους να σεβαστούν τον νόμο σου, ε, μπορείς να κάνεις πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα. Θα πρέπει να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι σχεδιασμένο για να αποτρέψει κάποιον ε, να προσαρτήσει παράνομα κάποια εδάφη. Θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και αποτελεσματικά που δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως είπα, επίση η διαφοροποίηση έχει καονιστική αξία. Γίνεται γιατί πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για να διατηρήσουμε και την ένωμη τάξη, του νόμου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικέ φορέ αναγκάζουμε το Ισραήλ να επιλέξει ανάμεσα στη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να συνεχίσει την ιδεολογική υποστήριξη των οικισμών. Όπως ακούσαμε τον ορίζοντα 2020, είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες στιγμές, ας πούμε, και σε προβληματισμούς πραγματικά ε, μοναδικούς και ενδιαφέροντες εντός του Ισραήλ. Ακόμα πιο σημαντικό είναι, σε μια στιγμή που υπάρχει μια τάση στο Ισραήλ να ε, εξομαλύνει, ας πούμε, και να ενσωματώσει τους οικισμούς, η διαφοροποίηση δεν θα σταματήσει την κατοχή, σε καμία περίπτωση αλλά παρόλα αυτά, αν εφαρμοστεί πλήρω είναι ένα φρένο σημαντικό στην, ε, στις τάσεις προσάρτησης του Ισραήλ. Έτσι, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους είναι προσάρτηση. Και τουλάχιστον διατηρεί την ε, Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη από αυτές τις διεθνείς παραβιάσεις και εξασφαλίζει ότι οι σχέσεις του Ισραήλ ε, με το Ισραήλ οι οποίες είναι απόλυτα θεμητές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υποσκάπτουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λύση των δύο κρατών. Ε, γιατί σε πολλές από τις διμερείς σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ το θέμα των οικισμών επισέρχεται. Επομένως, ε, δεν είναι ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαφοροποίηση. Υπάρχει και ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2016 το 234 για τη διαφοροποίηση και το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Ε, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κίνα πιο πρόσφατα, η Ιαπωνία πιο παλιά. Διάφορα κράτη συνειδητοποιούν ας πούμε το θέμα. Τώρα, τι μπορώ να προτείνω, τι συστάσεις μπορώ να κάνω. Να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαγγείλει μια αναθεώρηση των τρόπων ε, συμμετοχής ε, στην εξέβρεση λύσης των δύο κρατών. Το, το ανακοίνωσε η εκπρόσωπο εκπρόσωπο το Σεπτέμβριο. Εστιαζόμαστε στην οικονομική υποστήριξη προς το παρόν προς του Παλαιστίνιους. Ε, το θεμετό ερώτημα είναι αν αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να συμπεριλάβει και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Δεν σκοπεύουμε ούτε να τι περιορίσουμε σε καμία περίπτωση, ούτε να τι σταματήσουμε, αλλά τουλάχιστον δεν θέλουμε οι σχέσει αυτέ να μην ε, υποσκάπτουν τη θεώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λύση των δύο κρατών. Γι' αυτό λοιπόν ε, αποκλείουμε τις δραστηριότητες ε, των οικισμών από το πλαίσιο των σχέσεων με το Ισραήλ. Παράλληλα υπάρχουν και σχέσεις όμως ε, που έχουν τα κράτη-μέλη με το Ισραήλ. Δεν είναι μόνο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πέρα από τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δούμε τι κάνουν και τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει πρόοδος προς την κατεύθυνση της ε, διαφοροποίησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή η πρόοδος δεν υπάρχει στα κράτη-μέλη. Εμείς ε, έχουμε κατευθείαν γραμμέ χρηματοδότηση. Με την εξαίρεση τη ε, της Γερμανίας, κανένα άλλο κρατό μέλο δεν έχει κάνει το αντίστοιχο στο δικό του εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε. Ε, Επομένω, πρέπει να δούμε καταρχά τι κάνουν τα κράτη-μέλη στο δικό του εθνικό επίπεδο. Ε, υπάρχει η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με σκοπό την σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Ε, παρά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ε, παρά τον τεχνικ, τις τεχνικές διευθετήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι σχέσεις συμπεριλαμβάνουν τους, τα προϊόντα των οικισμών. Άρα ε, έχουν τις προτιμησιακές, ε, τους προτιμησιακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τα προϊόντα από, τα, ε, από τους οικισμούς. Επομένως, οι τεχνικές διευθετήσεις Ευρωπαϊκής Ένωση Ισραήλ ε, στρεβλώνουν λιγάκι την εικόνα ε, που πετυχαίνουμε τη διαφοροποίηση. Ε, και παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ε, αρμοδιότητε ε, στην εξωτερική πολιτική, επειδή έχετε αρμοδιότητε για την εμπορική πολιτική, μπορείτε να αντιμετωπίσετε μέσω αυτή αυτό το θέμα των τεχνικών διευθετήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ. Ευχαριστώ τον κύριο Πλόβατ. Ε, υπάρχουν ερωτήσεις ε, πρώτα. Λοιπόν, Άχιλα. Ε, ναι, καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω κουραστεί λίγο με τις δηλώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν μεταφράζονται ποτέ σε πράξη. Λόγια, λόγια, λόγια και τελικά δεν συμβαίνει τίποτα. 70 χρόνια διονύζεται η κατάσταση ε, εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εις βάρος της διεθνούς νομισμότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιτρέπει όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι την αλληλευτική συμφωνία που έγινε με το Μαρόκο, ε, για την οποία έγινε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί ε, χρησιμοποιούσαν τους πόρους της Σαχάρας σαν να ήταν πόροι του Μαρόκου. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν, ε, αφού θέλουμε να λάβουμε και άλλα σοβαρά μέτρα, να προσφύγουμε για αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ που στο άρθρο 2 λέει σαφέστατα το ότι αν δεν γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, θα ανασταλεί η συμφωνία. Γιατί λοιπόν να μην ε, προσφύγουμε στο δικαστήριο για αυτή τη συμφωνία. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά δεν θέλει να την αναστείλει, γιατί να μην προσφύγουμε εμεί στο δικαστήριο. Γιατί δεν τηρείται το άρθρο 2. Εγώ νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει άλλη λύση τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διεθνής νομιμότητα παραβιάζονται. Επομένως, το δικαστήριο λογικά πρέπει να αποφασίσει αυτό που πρέπει να αποφασίσει. Γιατί αυτό το μόνο που έχει ε, το Ισραήλ είναι αυτό το οικονομικό μοχλό πίεση. Ε, τα οικονομικά είναι και μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλέ άλλε πτυχέ ε, στα οποία θα μπορούσε να σταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αν θέλουμε να βοηθήσουμε να τηρείται η νομιμότητα και να είμαστε υπέρ τη λύση των δύο κρατών, πρέπει να γίνει σοβαρά. Ε, με εκπλήσει που λέτε εσείς όταν φτάσουμε σε ένα apartheid. Αν δεν είναι apartheid αυτό που ζούμε τώρα, ε, δεν ξέρω τι ε, αποκαλούμε apartheid. συνεχίζουμε να ε, συμπεριφερόμαστε στο Ισραήλ σαν να είναι μέλος της Ευρώπης. Eurovision, UEFA κλπ. Γιατί να την χάνει αυτή τη προνομιακή μεταχείριση. Από πότε είναι μέλος της Ευρώπης ε, το Ισραήλ. Εγώ δεν ξέρω γιατί του... Ε, ε αφιερώνουμε τέτοια συμπεριφορά, του, του συμπεριφορόμαστε με αυτόν τον τρόπο ε, να σας πω το εξή. Αν αυτό που κάνει ο νιάχου, το έκανε ο Μαδούρο ή οποιοδήποτε άλλος ε, πρόεδρος οποιασδήποτε άλλη χώρα ε, με αυτές τις οποίες έχουμε άλλες σχέσεις ή παίζουμε με άλλο τρόπο, να δούμε τι θα συνέβαινε, να δούμε ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι ε, ωραία και καλή διπλωματία και οι διεθνεί σχέσει, αλλά νομίζω ότι η υποκρισία περισσεύει πλέον σε αυτόν τον κόσμο, ιδίω όταν μιλάμε για ανθρώπου, τα δικαιώματά του και τη ζωή του. Διότι αν είμαστε τόσο υπέρμαχοι της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, το να καταδικάζουμε 70 χρόνια ένα λαό ο οποίος δεν έχει άλλη λύση και έχει μόνο να χάσει τη ζωή του, ουσιαστικά τους οδηγούμε στα άκρα και οποιαδήποτε λύση ε, δεν είναι σωστή για αυτούς. Ιδίω οι νέε γενιές ε, που εδώ και 70 χρόνια έχουν δει αντίσταση από το λαό τους για το τίποτα. Η διεθνής κοινότητα ε, κοιτάει από την άλλη πλευρά. αυτό συμβαίνει και 70 χρόνια εμείς είμαστε μάρτυρες αυτού. Τώρα, το BDS, το μποϊκοτάζ και τις κυρώσεις, λέτε ότι θέλετε. Όταν εφαρμόστηκε στην Νότια Αφρική ήταν νόμιμο και έδινε αποτελέσματα. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείτε ε, παράνομο κατά του Ισραήλ και θα πρέπει να μου το εξηγήσετε πάρα πολύ καλά. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν αρχίζει με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Γιατί δεν ξεκινάμε από εκεί. Για να δώσουμε ένα πραγματικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ήταν ένας τρόπος για να ξεκινήσουμε και να αποδείξουμε πραγματικά τη διάθεση για εξέβρεση λύσης και αναζήτηση λύσης σε αυτή τη διαμάχη. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και τέλος, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά ένα από τα μέτρα θα ήταν αυτή η συμφωνία να ε, αποτελέσει αντικείμενο προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, ευχαριστώ, αρχιλά. Ε, από και εγώ μερικά πράγματα ε, σαν ρωτήσω Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από αυτό που βάλε ο κ. Λόβατ για τα θέματα της ε, λύσης δύο κρατών και τη στάσεις στους Παλαιστινίους. Είναι αλήθεια ότι μέσα στην νέα γενιά των αυτό εισπράττουμε από τις επισκέψεις μας ε, τον τελευταίο καιρό στην Παλαιστίνη. Υπάρχει ισχυρή τάση ε, για να πάνε στην πολιτική ένα κράτος. Ε, και μάλιστα να πω ότι είναι αλήθεια ότι τη τελευταία συνεδρία του Παλαιστινιακού Εθνικού του Συμβουλίου της PLO, η οποία ανέδειξε την νέα ηγεσία, υπάρχουν όλο ένα και πιο περισσότερες φορές για να εγκαταλειφθεί η πολιτική ε, των δύο κρατών και να τερματιστεί η διαδικασία του Όσλου. Αυτό είναι ένα ε, νέο στοιχείο και διότι και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριο Λόβατο ότι ε, εάν πάνε σε αυτήν την λογική αυτό θα σημαίνει πόλεμος καθημερινός Δεν θα μιλούμε πλέον για ε, Θα μιλούμε για κάτι ίσως μια νέα αντιφάτα αλλά σε χειρότερη μορφή. Ε, και μπορώ να καταλάβω του ε, Παλαιστίνου. Τώρα για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ναι, συμφωνώ ότι θα γίνεται μια συζήτηση για την αναθεώρηση τη πολιτική, Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. το ότι κυρίω τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στη χρηματοδότηση. Ένα ζήτημα όμω που με προβληματίζει εμένα και αρκετού συναδέλφου, κύριε Λόβατ, όταν επισκεφτόμαστε την Παλαιστίνη, και πρέπει να σας πω ότι πηγαίνουμε τακτικά, θα έχουμε μια επόμενη επισκέψη το Σεπτέμβριο. Ε, αυτό που διεσάνομαι το τελευταίο διάστημα είναι μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να το θέλει, έμμεσα, αλλά με αυτή την πολιτική είναι σαν πως και χρησιμοποιητά την κατοχή. Η κατοχή χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Γιατί είναι κατοχική δύναμη το Ισραήλ. Είναι παντού ελέγχει τα πάντα και δεν έχει καμία υποχρέωση σε κάποιε πρόξει. Ούτε να λειτουργά νοσοκομεία, είτε σχολεία, είναι να χρηματοδοτά και όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει κατοχή ε, και ε, οι υπηρεσίε που προσφέρονται στου Παλαιστίνου, εκεί που είναι σε, κυρίως σε ε, area A, area B, ακόμα και area C που είναι οι, οι προσφυγικοί οικισμοί καμιά φορά, χρηματοδοτούνται οι περισσότερε υπηρεσίε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ε, και εγώ θεωρώ ότι το πρώτο ζήτημα είναι πρέπει να υπάρξει ε, αναγνώριση ε, και από τα κρατη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αναγνώριση δηλαδή του Παλαιστινιακού κράτου. Η πολιτική των δύο κρατών θα προχωρήσει στο βαθμό που θα μπορεί να αναγνωρίσει και να, να συμμετέχει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς παντού με το στάτους του κράτους το, ε, το, ε, το Παλαιστινιακό Στο βαθμό που θα υπάρχει αυτό το πράγμα, τότε θα είμαστε πιο κοντά στο να ε, ασκηθεί μια πίεση στο Ισραήλ για να προχωρήσει η πορεία ερνευση. Να πω την αλήθεια ότι εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο το μέρο που μα αναλογεί το έχουμε κάνει. Εμεί ω Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κράτη, αλλά το ότι. και ήταν μια εισηγήση δική μου τότε, τότε άλλαξε το όνομα τη αντιπροσωπεία από αντιπροσωπεία με το Παλαιστινιακό Ναστικό Συμβούλιο σε αντιπροσωπεία με την Παλαιστίνη, όπω γίνεται με όλα τα κράτη στο Κοινοβούλιο, αυτό ήταν, ένα, ε, ε, ήταν μια κίνηση που έριχνε ότι εμεί έχουμε, ε, έχουμε αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτο. Ε, Όμω είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται μια ευκαιρία, συμφωνώ με τον κύριο Λοβάτο, ότι έχει κάποια κόκκινε γραμμέ ε, που τι έθεσε και για την παραδοσία του Διεθνού δικαίου. Αλλά ε, θα πρέπει να κάνει περισσότερα από όσα κάνει. Και είναι ένα θέμα που και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να παρέμβουμε σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται για αναθεώρηση ε, τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχομαι στο τελευταίο μέρο που είναι το πιο ουσιαστικό σε σχέση με τη διαφοροποίηση. Ε, είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα. Ε, εγώ προσωπικά σε ό,τι αφορά την συμφωνία σύνδεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με το Ισραήλ. Έχω βάλει πάρα πολλέ φορέ θέση και στην Ολομέλεια ότι πρέπει να παγωποιηθεί αυτή η συμφωνία. Σαν μια κίνηση πίεση. Και πρέπει να, ε, να ε, παγωποιηθεί διότι το Ισραήλ παραβιάζει συστηματικά ένα βασικό άρθρο αυτής της συμφωνίας, το άρθρο 2, που είναι για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά και να παρακολουθούμε. Και το δεύτερο, ναι, μπορούμε να βάλουμε πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ σχέσει. Να πω ότι στην επέμονη επίσκεψη ε, στο Ισραήλ θα έχουμε καλέσει και πρόεδρου άλλων επιτροπών. Θα γίνει το Σεπτέμβριο από την Επιτροπή Εξωτερικών, από την Επιτροπή Πάτσετ και από την Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη να ε, συμμετέχουν οι προέδροι αυτών των επιτροπών μαζί μα στην αποστολή στην Παλαιστίνη σαν μια ευκαιρία να αποκτήσουν και γνώση και άλλες επιτροπές το τι γίνεται και ίσως ναι έχει εργαλεία να χρησιμοποιήσει κυρίως ό,τι αφορά το θέμα της διαφοροποίησης και το θέμα των εμπορικών σχέσεων το Κοινοβούλιο και, αλλά αυτό που θα ήθελα επειδή θέσετε αυτό το ζήτημα και σε σχέση με τη Συμφωνία Ελευθερών Πορείου εάν μπορείτε κύριε ε, Λόβα να μας πείτε ε, Δύο λόγια περισσότερο. Δηλαδή, ποιο θα μπορούσε να ήταν το επόμενο βήμα σε σχέση. Ε, ένα στοιχείο έχουμε αυτό που έγινε και με το ορίζοντα 2020 και με τα θέματα ε, των προϊόντων από οικισμού, αλλά τι είναι το επόμενο βήμα που θα μπορούσε να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση και από πλευρά Κοινοβουλίου για να μπορεί να ασκηθεί μια μεγαλύτερη πίεση. Ο Ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι η πρώτη παρατήρηση, και αυτό εννοούσα όταν ξεκίνησα με τα προκαταρκτικά μου σχόλια για την ε, ε, λύση των δύο κρατών και τις συνέπειες. Σίγουρα θα υπάρχουν βαθιές συνέπειες για το Ισραήλ και βαθιές συνέπειες για τους Παλαιστινίους, αλλά επίσης ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους Ευρωπαίους. Και νομίζω ότι αυτό τους επηρεάζει αρκετά και οι Ευρωπαίοι θεωρούν, ε, σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία, ότι είναι υπερασπιστές του status quo ε, και ε, επιτόπου και στο διεθνέ προσκήνιο. Και πρέπει περιττό να πούμε ότι το status quo επιτόπου είναι ένα λαθασμένο status quo και αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση οτιδήποτε μπορεί να προηθήσει και είναι θετικό, ε, ξεπερνιέται από τις εξελίξεις επιτόπου. Το διεθνέ status quo παραμένει ω τι τελικέ θέσει ε, και τι αποφάσει. Ε, και τη αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται διεθνώ, αλλά υπάρχουν και δράσει από την ε, ε, Αμερικανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, την κυβέρνηση Τραμπ, για τι οποίε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει. Αυτά τα οποία γίνονται και επί τόπου και διεθνώ είναι το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε τις σχέσεις μα με την PLO αλλά και με το Ισραήλ. Ε, τις συμφωνίες σύνδεσης. Πώς ερμηνεύονται αυτά σε μια κατάσταση στην οποία επιθετικά στο μέλλον δεν θα υπάρχει ε, πλέον ε, η λύση των δύο κρατών, θα έχει εξαφανιστεί, θα θεωρείται ότι είναι κάτι ανέφικτο και θα δεχτούν όλοι ότι αυτή είναι η κατάσταση apartheid. Πώς θα ερμηνεύουν τη συμφωνία σύνδεσης και τις υπόλοιπες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και η PLO θα πρέπει να κάνει κάτι το οποίο να μπορέσει να πείσει από πολιτική σκοπιά. Ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι ε, προϊόντα αναστολή της συμφωνίας επειδή έχει αλλάξει, αν αλλάξει μάλλον η κατάσταση και βρεθούμε κάπου μετά από τη λύση των δύο κρατών, θα είναι πολύ δύσκολο η Ισραηλινή κυβέρνηση να ε, αιτιολογήσει γιατί δεν κάνει κάποια πράγματα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι θέλει να βγάλει τους Παλαιστινίους εκτός ε, διαπραγματευτικού τραπεζιού και αν τα καταφέρουν φυσικά θα υπάρχουν συνέπειες για το Ισραήλ στο μέλλον γιατί αυτό θα αλλάξει και την ουσία των σχέσεών του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια σε αυτό το σημείο ακόμα και ακόμα προς το παρόν έχουμε αυτό το μοντέλο ε, ειρήνευσης με λύση των δύο κρατών. Και νομίζω ότι είναι πολύ πιο τραγικό ότι υπάρχει μια Παλαιστινιακή πλευρά με τα πολλά ασφάλματα, ε, την Παλαιστινιακή ηγεσία ε, και δεν το λέμε για να τους ε, ε αθώσουμε για κάποια πράγματα στους Παλαιστινίους, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παρά τα πολλά του ε, ε, ελαττώματα, ο Αμπάς είναι πεπισμένος για τη λύση των δύο κρατών, παρά τα όσα κάνει ε, είναι πεπισμένος ότι πρέπει να προχωρήσουν οι συμφωνίες του Όσλο και συντονισμό σε θέματα ασφαλείας με το Ισραήλ δηλαδή, και επίσης παρά ρητορικές που φορές είναι και τις παραφές ε, της, ε, του αντισημιτισμού ή και σαφώς αντισημιτική, βλέπουμε από τις ε, πράξεις του ότι είναι υπέρμαχος της λύσης χωρίς βία για την στρατηγική απελευθέρωση απελευθέρωσης Παλαιστίνης. Και όλα αυτά τα λέω γιατί Υπάρχουν πολλές επικρίσεις για τον Αμπάς, αλλά νομίζω ότι ήταν ένας από τους πυλώνες του παρόντος μοντέλου της ειρηνευτικής διαδικασίας. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί μετά από αυτόν. Υπάρχουν αρκετές προκλήσεις και δυναμικές ε, και από την Παλαιστινιακή πλευρά που θα αμβληθούν. Ιδιαίτερα ε, καθώς οι νέες γενές Παλαιστινίων θα αρχίσουν να αποκτούν εξουσία σε 10-15 χρόνια άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μετά από τις συμφωνίες του Όσλο, που ε, ήταν πολύ νέοι για την πρώτη Ιντιφάντα ε, και, και δεν είχαν γεννηθεί μάλλον στην πρώτη και ήταν πολύ νέοι στη δεύτερη. Και η λύση δεν θα είναι μία χώρα ή δύο χώρες, θα είναι ισότητα, αξιοπρέπεια, ακόμα και υποκατοχή. Και επομένως θα πρέπει να δουν πώς θα διαρθρώσουν την πολιτική τους για τη στρατηγική τους και θα είναι λίγο διαφορετική από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι τις παρούσεις, είναι μελλοντικά. Και νομίζω, όπως σας είπα, ότι το ερώτημα είναι αν μπορεί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Νομίζω ναι, αλλά το θέμα είναι θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα καταφέρει και να ε, υπάρξει και η πολιτική βούληση. Δεν είναι μόνο ότι η Γάζα, η ζώνη Γάμα, οι κατεδαφίσεις κλπ θα είναι προετοιμασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα κάνει όλα αυτά και να δει και τους εσωτερικούς τους κανόνες να λειτουργούν όπως πρέπει και να μην παρεμβαίνει για πολιτικούς σκοπού για να προλάβει ε, τη μη σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό γι' αυτό. Αν γίνονται κάποια πράγματα, ορισμένε φορέ γίνονται ad hoc, γίνονται με πολύ αργά και τα ξεπερνούν οι αρνητικέ εξελίξει. Το μόνο πράγμα που θα αλλάξει τα πράγματα είναι αν υπάρξει μια συνολική αποδοχή ότι πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι καλό και πρέπει να γίνει και κάτι καλό θα κάνει εάν συμβεί. Και αυτό δεν θα αφορά μόνο το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πρέπει να πάμε και σε επίπεδο κρατών μελών και ούτω καθεξής. Και δεν αφορά μόνο να πάμε σε νέες τομεί, γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι τομεί οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ε, φυγεί. Ε, τα οικονομικά, για παράδειγμα, είναι πολύ περίπλοκα Υπάρχει το θέμα της ενέργειας, πολλά τεχνικά ζητήματα, αλλά αφορά και την εφαρμογή ε, προηγούμενων συμφωνιών για τις εμπορικές συμφωνίες ε, σχέσεις με το Ισραήλ, για την ε, επισήμανση στα προϊόντα. Υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές, αλλά σε μεγάλο βαθμό δεν εφαρμόζονται. Αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν το παιχνίδι μεμονωμένα, αλλά εάν γίνουν με πιο ολιστικό ε, και συντονισμένο τρόπο, τουλάχιστον θα ε, αποτελέσουν και μία πρόκληση και οι προσπάθειες της Ισραηλινής κυβέρνησης και των επικασμών να υποσκάψουν το διεθνές δίκαιο και να επιβάλλουν τη δική τους θέση, η πράσινη γραμμή που εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική λύση για τη λύση των δύο κρατών. Και όσον αφορά την αναγνώριση, νομίζω ότι η επιτυχία των γαλλικών κυβερνήσεων και ο Λαντ και ο Μακρόν είναι ότι έθεσαν δύο προϋποθέσεις για την αναγνώριση. Κατάλληλη χρονική συγκυρία και τι αντίκτυπο θα έχουν. Πότε θα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή και τι αντίκτυπο θα έχει. Όσον αφορά τη χρονική συγκυρία, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν είναι τώρα η καλύτερη στιγμή, δεδομένες και της κατάστασης επιτόπου και το θέμα του αν θα επιβιώσει η λύση των δύο κρατών. Για να μην σας πω ότι είναι και πολύ αργά, αν φανώ πολύ απεσιόδοξος, ε, αλλά ναι, μεν όλοι συζητούν τη λύση για τον δύο κρατών και μένουν μόνο δύο χρόνια και έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και ακόμα συζητάμε για το ίδιο θέμα. Αλλά μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τι προκλήσει για μια λύση δύο κρατών. Είναι πολύ συγκεκριμένε και νομίζω ότι η αναγνώριση είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα ζωή στη λύση των δύο κρατών. Μπορεί εν τέλει να μην χρεια... αρκέσει, αλλά όσον αφορά τον αντίκτυπο και το συμβολισμό, κάτι προσφέρει και υπάρχουν και συνέπειες σε διεθνέ δίκαιο για τον τρόπο με τον αντιμετωπίζουμε του Παλαιστινίου και ότι θα πρέπει να περιμένουμε και από το Ισραήλ ε, και δική μας διαφοροποίηση. Και θεωρώ ότι αυτά ε, αποτελούν σωστή απάντηση και αν ρωτήσουμε και τα κράτη-μέλη πώς αιτιολογούν να μην κάνουν τίποτα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λοβάκ. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για σήμερα. Α, στα διάφορα δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση. Ε, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να πω ότι η επόμενη συνεδρία θα γίνει στο Στρασβούργο 4 Ιουλίου από τις 3 μέχρι τις 4.30. Ε, θα σταλεί από τη Γραμματεία η ημερήσια δίδαξη και λεπτομέρειε. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και ευχαριστώ τους διερμηνείς για την συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίας μας. Ευχαριστώ.